So we will start to vote. And now... Ωραία λοιπόν, περνάμε στο σημείο 6 της σημερινής σας διάταξης, οι υπηρεσίες οικονομικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων. Η συνάδελφος Σύρπα Πιτικάινεν είναι η συγκεκριά μας και έχουμε μπροστά μας την υιοθέτηση του σχεδίου της έκθεσης. Ε, τροπολογία 1-2-2 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 123 σε δύο ε, τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 124. 124. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 125 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία θέλετε να ελέγξετε την 125. Καλώς ελέγχουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία την 125. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 126 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ Sorry, sorry. 126. 126. Τροπολογία 126. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 127 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Καλώς ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα της 127 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίες Εγκρίνεται. 127 πάντοτε. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 135 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 135. Αρχιτεί ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 136. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 137 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε την τοπολογία 137. Άρχεται η ψηφοφορία. Τώρα λοιπόν ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 138 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 249 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 153 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 166, 167 και 168 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τροπολογία 176 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 179 σε τρία τμήματα υπέρ όχι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 186 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 187 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 188 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 189 υπέρ 192 συγγνώμη υπέρ κατά εποχές να την ε, ελέγξουμε την 192 ελέγχουμε την 192 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εκρίνεται. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 17 υπέρ. Συμβαστική τροπολογία 17 υπέρ. Κατά αποχές ας ελέγξουμε τη συμβαστική τροπολογία 17 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 204 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 205 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 203 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 207 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 200 208 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 209 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 217 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 219 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 233 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 200 234 και 235 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 236 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 215 και 273 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται συμβαστική τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 241 και 242 υπέρ κατά 241 και 242 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2. Ναι, μπορούμε να ελέγξουμε λοιπόν τις 241 και 242 άρχεται η ψηφοφορία. πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτονται. 2.43 υπέρ, κατά Επαναλαμβάνω, 2.43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να την ελέγξουμε. Ωραία. Ελέγχουμε τη 2.43 ηλεκτρονικά, έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 244 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 2.52 υπέρ κατά αποχές εκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 278 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 253 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 251 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 283 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 287 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 200 84 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 286 υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε την 286, ε, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρασε της ψηφοφορίας. Amendment 288. 288 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 289 υπέρ. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 290, 291, 294 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. άποχε, Εγκρίνονται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές Ας ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. And now the vote is closed. It... Εγκρίνεται. Uh, amendment 292 in two... Η δεις. σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, παρακαλώ. Ε, η κάρτα μου, η κάρτα μου. Είναι στην Επιτροπή Γιούρι. Τώρα μου τη φέρνουν. Δεν μπορώ να ψηφίσω με την κάρτα.

Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μπορούμε να καταμετρήσουμε την ψήφο σας, λέει η Πρόεδρος. Μπορούμε να ψηφίσουμε, να καταμετρήσουμε την ψήφο σας, μόνο εάν δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση αλλάζει το αποτέλεσμα. Στην Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων, όταν δεν έχω την κάρτα, με αφήνουν να ψηφίσω. Και είναι Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Το λέω μήπως και άλλαξε τους κανόνες. Which now, which now we, we need... Uh, we need... 290. Okay. Second part, 290. Aha. 90, Dear colleagues, Συνάδελφοι. Which part? Which ah. Ah, Συνάδελφοι, 290-291 καταπίπτουν. Το δεύτερο τμήμα θα το ψηφίσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Vote Ψηφίζουμε. Και πέρασε. Απορρίπτεται. Η 2.92 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 302 υπέρ. Κατά. 302. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 305 και 306. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 311. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 312. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχο ζητείτε για τον συμβαστική 3. Εντάξει λοιπόν. Έλεγχο. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τη συμβαστική υπαριθμό 3. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 56 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Σεμιβαστική 4 για την 57 ελέγχουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Και πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ Θέλετε να ελέγξουμε την 70 Εντάξει, ελέγχουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 70 ψηφίζουμε και πέρας Απορρίφθηκε. Η 73 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 81 και 82 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Έλεγχος για την 81-82. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Α, καταπίπτει. Η 85. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 1, 3 και 14 από κοινού υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8, 9 και 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13, 15, 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όλες ναι μαζί από κοινού. Οι 13, 15 και 17 είναι ταυτόσημες. Και ως εξουστούνται τις ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Οι 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 και 26 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. έγκρίνεται. 34 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 θέλετε να ελέγξουμε παρακαλώ 31 εντάξει ψηφίζουμε την 31 όχι δεν θέλετε να γίνει έλεγχος ψηφίζουμε ψηφίζουμε πέρας ψηφορίες τώρα εγκρίνεται η 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα με ηλεκτρονική ψηφοφορία το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Και πέρας. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια στην κυρία Πιετικά είναι την εισηγήτρια και ευχαριστούμε επίσης όλους τους κοιόδες. Και στη Λέα, συγχαρητήρια. Και τώρα πάμε στο 7. Έχουμε την ε, ενδιάμεση έκθεση για τα έτη 2021-2027, η θέση του Κοινοβουλίου εν ώψη της ε, συμφωνίας. Η εισηγητής, η εισηγήτρια μάλλον κυρία Ράτσεγκαρθία Πέρεθ και έχουμε τώρα την ψήφιση ε, αυτού του σχεδίου κειμένου και των τροπολογιών. Η 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 σε δύο τμήματα το πρώτο τμήμα Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο. Μάλιστα. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφορία. Και εγκρίνεται. Ε, which now, which are Uh, amendment 27 in favor.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 για το πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρα της Να σηκώνετε τα χέρια σας. Και τώρα. Για το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, να κάνουμε έλεγχο. Τρίτο τμήμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος. ψηφίσμου, Και τώρα πέρας της ψηφορίας. Και εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Ναι.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 και εγκρίνεται. Συγχαρητήρια, κυρία Ιράτσε. Και συγχαρητήρια σε όλους τους σκιώδες ηγητές που συνεργάστηκαν. Point on the agenda. Κοινέ διατάξεις, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και τα λοιπά και τα άλλα ταμεία. Τζούλι Γκέρλινγκ είναι η εισηγήτρια. Έγκριση και διοικημένου κειμένου κοινή θέση και των τροπολογιών. Ξεκινούμε. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 σε δύο τμήματα. Το πρώτο υπέρ. Καταπίπτει λέει η γραμματείας. Α, μάλιστα λέει πρόεδρος. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε για το 18 το πρώτο τμήμα γιατί καταπίπτει. in favor. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19. Εις δύο τμήματα το πρώτο. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. 20 σε δύο τμήματα το πρώτο. Υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται.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 εγκρίνεται να κάνουμε έλεγχο στο δεύτερο τμήμα, όπως θέλετε. Ψηφίζουμε. Και τώρα είναι το πρέσβη ψηφορίας και εγκρίνεται. 37, υπέρ κατά, εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46 σε δύο τμήματα. Για το πρώτο. Υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίντε. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχε εγκρίνεται. 48 σε δύο τμήματα υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται το πρώτο μέρος. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται.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 No. The first part falls and the second part... Ah, recital, yeah. Recital Πρώτη του λογική. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα, 7. Σε δύο τμήματα. Το πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 11. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και η 13. Υπέρ κατά και αυτή εγκρίνεται. Ευχαριστούμε. Μπράβο στην Τζουντιγκέλη και του και τους nine uh, the situation of women with disabilities. Reporter, uh, uh, Ms. Rosa. Ε, περνάμε στο σημείο 9 ε, της σημερινής διάταξης, ε, των γυναικών με αναπηρία. Ε, με εξηγήτρια την ε, κυρία Στέρα Φραγκούτ. Και περνάμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ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 23 υπέρ κατά αποχές πρέπει να την ελέγξουμε. Την 23 υπέρ, ε, συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 Να ελέγξουμε την 26 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 29 σε τρία τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα λοιπόν της 31, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τριάντα δύο υπέρ. Κατά αποχές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 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικά. Ωραία, τη 48 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 50 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά αποχές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 κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 σε 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 10 σε δύο τμήματα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην ε, τελική ψηφοφορία για το σχέδιο της έκθεσης σχέδιο μάλλον ψηφίσματος ε, έτσι όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. Συγχαίρουμε λοιπόν την εισηγήτρια, την κυρία Ρόζα Σταράς Φεραγκού. we don't need to vote on this is the cover. No. No. This no. one. This one. Aha. uh -huh. And now. Uh, the, There are two requests for the floor. Yes, please. Uh, yes, Ms. Zaborska, please. Yes. Uh, merci, Madame la Présidente. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να καταθέσω την ε, άποψη της μειονότητας σε ό,τι αφορά την έκθεση που μόλις ψηφίσαμε. minority position. And this file. For me. You, you need to ask. Sorry. Yes, please. I ask, this, I ask the same as Madam Zaborska. Και εγώ το ίδιο ζητώ, όπως η κυρία Ζαμπόρσκα, τοποθέτηση της μειοψηφίας. Ναι, φυσικά, μετά την ε, ψηφοφορία όμως, λέει η Πρόεδρος. Um, Προφορική ερώτηση για την κατάσταση των γυναικών με αναπηρία. Το κείμενο στο σύνολό του ψηφίζουμε, παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Ηλεκτρονικά, λέει η Πρόεδρος. Την προφορική ερώτηση, παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Everybody's vote now. Ψηφίστε παρακαλώ όλοι. Πέρας. Όχι, μας λείπει ένας ακόμα. I think we can close. And the vote now is closed. Okay, Πέρας. Μάλιστα. Εγκρίθηκε συγχαρητήρια.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 Συνάδελφοι, στο σημείο 10 της ημερησία διάταξη έχουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για δράσεις για τα κορίτσια. Ανταλλαγή απόψεων με δύο εκπροσώπους των νεαρών γυναικών και θα μας παρουσιάσουν και κάποιες βασικές συστάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και για την εξασφάλιση της δέσμευσης τους για τον αγώνα για τα δικαιώματα των κοριτσιών και μετά ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να σας ενημερώσω δε ότι η συνεδρίαση άμα θα καταγραφεί. Έχουμε κάποιον που παίρνει βίντεο και θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην Χάμντι Άριφ, η οποία είναι πρέσβης της νεολαίας και ακτιβίστριας με την Ομοσπονδία των Ενώσεων Σομαλίας στις κατοχώρες FSAN. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Λειτουργεί το μικρόφωνο μου. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν. Ονομάζομαι Χάμντι Αρίφ και καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους εσάς ε, τους ευρωβουλευτές που σήμερα μας ακούτε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που συνεχίζετε να ακούτε τις φωνές της νεολαίας και θα ήθελα όλος ο ιδιαίτερος να σας ευχαριστήσω για την συνεχιζόμενη διαδημευσή σας για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών και ε, παρακολουθούμε τις εργασίες της Επιτροπής σας τα τελευταία πέντε χρόνια. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την τήρηση των υποσχεσεών σας και για το γεγονός ότι δεν ξεχνάτε ποτέ τι έχει σημασία για τις νεαρές γυναίκες και για τα κορίτσια. Νομίζω ότι μιλάω εξ ονόματος όλων των κοριτσιών όταν λέω ότι οι πολιτικοί θύνοντες όπως εσείς που ε, εξασφαλίζουν ότι οι πολιτικές ε, και οι επενδύσεις ε, έχουν τα αποτελέσματα που χρειάζεται στη ζωή μας και πάνω απ' όλα που εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματά μας κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική για μας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι. Βρισκόμαστε σήμερα στην αίθουσα αυτή από διάφορες χώρες, από διάφορα, πολιτικά υπόβαθρα, γιατί μας ανώνει ένα κοινό όραμα Θέλουμε ένα κόσμο όπου όλες οι γυναίκες, όλα τα κορίτσια ζουν ελεύθερα, ευτυχισμένα, με την ε, δύναμη που τους αναλογεί. Και για τον λόγο αυτό λοιπόν τα Ηνωμένα Έθνη αποφάσισαν να αφιερώσουν μια ημέρα την 11η Οκτωβρίου στις, ε, στα κορίτσια. Δυστυχώς. Το 2018, λίγο πριν την διεθνή αυτή ημέρα, η ικανοποίηση και η ευτυχία απέχει ακόμα πολύ από, την, ε, από πολλές γυναίκες και παιδιά. Είναι τραγικά τα ποσοστά των γυναικών που παντρεύονται καταναγκαστικά πριν το 18ο χρόνο τους. Ε, αυτό σημαίνει και λιγότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη, καριέρα και με πιο πολλές ε, πιθανότητες για ενδοοικογενειακή βία. Κυρίως και τουλάχιστον 200 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες ε, σήμερα έχουν υποστεί ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων με ό,τι αυτό συνεπάγεται ψυχολογικά και σωματικά. Στις πιο πολλές χώρες ε, αυτό γίνεται πριν από την ηλικία των 15 χρονών. Και αυτό δεν είναι θέμα που αφορά μόνο την Αφρική. Στην Ευρώπη μόνο οι γυναίκες και τα κορίτσια άμα και γυναίκες που έχουν υποστεί ακροτηριασμό γεννητικών οργάνων υπολογίζονται σε 500.000 στην Ευρώπη. Και μεγάλο είναι το ποσοστό γυναικών που έχουν υποστεί ψυχολογική ή σωματική βία. Αυτή η βία επηρεάζει οι νεαρές γυναίκες όπως και εγώ. Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί τέτοια βία πριν την ηλικία των 15 από ενήλικους και δυστυχώς αυτά τα αριθμητικά στοιχεία θα μπορούσα να συνεχίσω να σας τα παραθέτω. Δεν ήλθα όμως εδώ σήμερα ενώπιον σας για να μας ε, κάνω όλου ε, να θυμώσουμε. Εγώ είμαι Ολλανδή, από τη Σομαλία είναι η οικογένειά μου και ο ακροτηριασμός ε, γεννητικών οργάνων είναι μια πρακτική που πλήττει 95% των γυναικών, συμπεριλαμβανομένη και τη μητέρα μου, η οποία αγωνίζεται εδώ και 25 χρόνια κατά τη πρακτική είπε ότι φτάνει πια. Η κόρη τη ε, δεν θα υπόκεινταν την ίδια ακροτηριασμό. Θεωρώ ότι είμαι τυχερή γιατί η μητέρα μου με προστάτευσε και εμένα και τι αδερφές μου. Είναι με πραγματική έμπνευση. Και έχω αφιερώσει την ε, ζωή μου στην ε, καταπολέμηση αυτής της πρακτικής από την οποία γλίτωσα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προωθήσουμε και το δικτυό μας, το NFGM και γι' αυτό βρίσκομαι λοιπόν εδώ σήμερα. Έχετε λοιπόν ως Ευρωκοινοβούλιο ε, βασική αρμοδιότητα και μπορείτε να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο στη ζωή εκατομμυρίων κοριτσιών στον κόσμο. Ζητάμε λοιπόν μια αποτελεσματική στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να καταπολεμηθεί οποιαδήποτε διάκριση και βία κατά των κοριτσιών και στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό θα πρέπει να γίνει λοιπόν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δαπανίσει και να επενδύσει σε προγράμματα ευαισθητοποίησης όχι μόνο για γυναίκες και κορίτσια αλλά και κοινότητες όπως αυτές των ανδρών και των ηγετών θρησκευτικών κοινοτήτων. Αυτό επηρεάζει και όλες τις μορφές βίας στον κόσμο σε ό,τι αφορά τη συνεργασία για την ανάπτυξη και να καταδικάσει και να εντάξει την ρεσιμότητα για την ενδοκογενειακή βία στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. καθημερινά θα πρέπει να πολεμήσουμε τέτοιου είδους ε, μορφές βίας ε, γιατί δάλλως θα συνεχίσουν τα πράγματα όσα έχουν και θα χάσουμε τη φωνή μας σε μια κοινωνία και έτσι θα παραβλεφθούν τα δικαιώματά μας και οι ανάγκες μας. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πρωταθλήτρια για τα κορίτσια και για τις γυναίκες και να προωθήσει την πολιτική ενδυνάμωσης προκειμένου να προσθεθούν και όποια προγράμματα ενδεχομένω βοηθήσουν τι γυναίκε. Με ίση εκπροσώπηση των γυναικών. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί με τρίτε χώρε για να έχει πιο καλή συνεργασία με του νέου, για να υπάρχει μια ανοιχτό πνεύμα και μεγαλύτερη συμμετοχή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρί τι απαραίτητε ε, επενδύσει, τον απαραίτητο προπολογισμό. Γι' αυτό λοιπόν στην παρούσα φάση είναι απαραίτητο εσείς ως ε, βουλευτές να ζητήσετε ένα νέο οικονομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έχει στην επίκεντρο την νεολαία. Συμμετοχική λοιπόν και κοινοτομική προσέγγιση προς τους νέους και κυρίως προς τις γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια. Είναι επίσης ε, απαραίτητο να υπάρχει ευελιξία στη χρηματοδότηση προκειμένου να μπορούν να διαχειρίζονται τους πόρους αυτούς ε, οι τοπικές ενώσεις ακτιβιστριών. Μόνο έτσι θα πετύχουμε πραγματική αλλαγή. Μέσω της συμμετοχής των κοριτσιών και της ενδυνάμωσης των κοριτσιών και μόνο με τον τρόπο αυτό θα πετύχουμε να ξεπεράσουμε τη βία και πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε. Καλή Παγκόσμια ημέρα κοριτσιών και γυναικών και ελπίζω αυτό να είναι η αρχή και μόνο μια συγκεκριμένη δράση που θα έχει αντεκτύπω για κάθε γυναίκα και κάθε κορίτσι. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Ms. Kandi Arif. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Κάντι Αρεπ. Και δίνω τώρα τον ε, λόγο στην κυρία Φελίστια Σεμπέργκερ ε, πρέσβυρα της νεολαίας και επικεφαλής του Euro Foundation ε, στον τομέα της ηθικής αριστείας. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την αδερφή Χαμντή ε, για την εισαγωγή που έκανα. Θα ήθελα να αλλάξω αυτή την ευκαιρία Σε αυτήν εδώ λοιπόν, το, σε αυτό το κοινοβούλιο ε, συζητούνται σημαντικά ζητήματα καθημερινά και κατά συνέπεια είναι δική μου υποχρέωση ω πρέσβυρα τη νεολαία να μεταφέρω τι φωνέ τη νεολαία σε εσά εδώ. Ε, πριν από μερικά χρόνια είχα τη δυνατότητα να εργαστώ και να ζήσω στο Καμερούν και ήμουν τόσο εντυπωσιασμένη με τον τρόπο που τα κορίτσια και οι γυναίκε εκεί αντιμετωπίζουν τι καθημερινέ δυσκολίε τη ζωή. Ε, ε Σκεπτόμενο δηλαδή το σχολείο, εργαζόμενο ε, ε, και μαγειρεύοντα για το σπίτι. Ουσιαστικά δηλαδή δεν είχαν σχεδόν καθόλου χρόνο στη διάθεσή τους για να κάνουν ε, όσα είχαν να κάνουν για το σχολείο στο σπίτι τους και αυτό βέβαια ε, συνέβαινε μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου ε, δεν τις έβγαζαν οι γονείς από το σχολείο έτσι ώστε να εργάζονται μόνο στο σπίτι. Άρα λοιπόν διαπίστωσα πόσα πολλά ταλέντα χάνονται εκεί ακριβώς επειδή τα κορίτσια δεν έχουν δυνατότητες στη διάθεσή τους, δεν έχουν ευκαιρίες. Άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτά τα κορίτσια και να κάνουμε την αλλαγή έτσι ώστε να ε, ε, να μην επιτρέψουμε το να μεγαλώνουν τόσο γρήγορα, τόσο πρόημα και να τις ε, επιτρέψουμε να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Και γι' αυτό λοιπόν έγινα και εγώ πρέσβα της νεολαίας έτσι ώστε να υψώσω τη φωνή μου για αυτά τα κορίτσια και τις γυναίκες που γνώρισα στο Καμερούν. Εγώ είχα την τύχη να μεγαλώσω στη Γερμανία. Είχα λοιπόν μια ασφαλή οικία, μια καλή εκπαίδευση και στην ηλικία των 24 έχω ακόμα τη δυνατότητα να σπουδάζω για να γίνω ιατρός θέλω να έχω μια καριέρα ε, σε αντίθεση με την ε, μητέρα μου η οποία χρειάστηκε να αναθρέψει εμένα και τα αδέρφια μου ενώ ο πατέρας μου ε, δούλευε. Και αυτό παρότι η μητέρα μου είχε περισσότερες δεξιότητες και το λυπηρό αληθέ είναι ότι ακόμα και αν εργαζόταν εκείνη με τι περισσότερε δεξιότητε, θα έβγαζε λιγότερα χρήματα από ότι ο πατέρα μου. Και αυτό είναι αποδεκτό σε μια χώρα όπω η Γερμανία, η οποία θεωρείται ω μια από τι πιο ανεπτυγμένε στον κόσμο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να αποδεχόμαστε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να δείξουμε στα κορίτσια ότι είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν τα όνειρά του με τον τρόπο που τα πραγματοποιούμε εμεί. Δεν θα πρέπει να υπάρχει τίποτα που να τα εμποδίζει. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία χώρα σε αυτόν τον κόσμο, ούτε μία χώρα όπου οι γυναίκε έχουν τι ίδιε ευκαιρίε με του άντρε. Δεν υπάρχει ούτε μία χώρα όπου να συμβαίνει αυτό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το να γεννιέται κανεί γυναίκα, πέρα του να γεννιέται φτωχή, είναι ουσιαστικά ένα διπλό βάρο. Ένα διπλό άχθο. Και θα ήθελα να, σε αυτό το πλαίσιο να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη εδώ αυτή τη Επιτροπή ΦΕΜ, έτσι ώστε να σα παρουσιάσουμε την κατάσταση αυτών των κοριτσιών, προκειμένου να βελτιώσουμε τι ευκαιρίε των κοριτσιών ανά τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω γνωρίζετε, έχει ήδη αναλάβει μία σειρά από δεσμεύσει. Υπάρχει η ατζέντα του θεματολόγιου του 2030 σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Συμφωνία για την Ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Σχέδιο Δράση του Ντένβερ, η Πρωτοβουλία ε, Spotlight και η Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανταποκρίνεται στι υποχρεώσει, στι δεσμεύσει που έχει αναλάβει στο πλαίσιο όλων αυτών των συμφωνιών. Ούτε τουλάχιστον δεν το κάνει ακόμα. Είναι ε, σημαντικό λοιπόν να ε, ταχθεί, ε, θα πρέπει να ταχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ των κοριτσιών. Αυτό σημαίνει δηλαδή να προωθήσει περισσότερο την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και να ε, αποτρέψει ε, για να καταπολεμήσει τι διακρίσει σε όλο τον κόσμο. Τώρα με τι επικίνδυνε ευρωπαϊκέ εκλογέ νομίζω πω είναι κατάλληλη ευκαιρία ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δείξει ότι βρίσκεται στο πλευρό των γυναικών και των κοριτσιών ανά τον κόσμο. Εσεί ω μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να δείξετε ότι τα δικαιώματα ε, των κοριτσιών και των αρρών γυναικών λαμβάνονται πόντοτε υπόψη σε όλε τι δράσει του Κοινοβουλίου. Οι ευρωβουλευτέ μα και θα πρέπει να διασφαλίσουν επενδύσεις οι οποίες εξασφαλίζουν περισσότερες ευκαιρίες για αυτές τις γυναίκες. Και πιστεύουμε ότι το 85% των κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να κατευθύνονται σε project τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους στη διάσταση του φύλου. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή την περίοδο συζητάται ο επόμενος μακροπρόθεσμος, μακροχρόνιος προπολογισμό της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και του Κοινοβουλίου. Ε, πέραν λοιπόν αυτού θα πρέπει το Κοινοβουλίο να δώσει περισσότερη έμφαση στα ζητήματα τα οποία απασχολούν περισσότερο τι γυναίκε, ειδικότερα σε ό,τι αφορά δηλαδή την ε, απόδοση αυτεξουσιότητα ε, σε αυτές και τη συμμετοχή στα κοινά. Θα πρέπει να σταματήσουμε κάθε είδους δυσμενείς διακρίσεις και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η οικονομική αυτάρια και η δυνατότητα εκπαίδευσης να αποτελέσουν πραγματικότητα για όλες τις γυναίκες. Ε, τι σημαίνει όμως empowerment, απόδοση αυτοεξουσιότητα, Σημαίνει ίσες ευκαιρίες για όλους παντού. Σημαίνει το να μπορούμε να ε, πραγματοποιούμε το πλήρες μας δυναμικό. Πράγμα το οποίο ξεκινά από τις πρώτες ημέρες της ζωής μας. Και κατά τη δική μου άποψη όλα ξεκινούν από την ε, παιδεία. Εγώ είχα τη δυνατότητα να σπουδάσω, να μάθω διάφορα πράγματα και να έχω διάφορες εμπειρίες ε, στη ζωή μου και θεωρώ πως πραγματικά η παιδεία είναι ε, το σημαντικότερο εργαλείο με το οποίο μπορούμε να ε, επιτύχουμε περισσότερη αυτοξουσία για τις γυναίκες. Και εδώ έχω και κάποια ενδιαφέρουσα, ενδιαφέροντα δεδομένα. Για παράδειγμα, μία φίλη μου η οποία επισκέπτεται το σχολείο στο Καμερούν με κάθε παραπάνω έτος μπορεί να αυξήσει κατά 12% το μισθό της. Ενώ ε, μία τέτοια αύξηση του παιδιού ζωής θα μπορούσε να βοηθήσει στο να σωθούν 1,2 εκατομμύρια ζωές ε, παιδιών. Παρόλα αυτά ε, έχουμε τη σήμερα 130 εκατομμύρια κορίτσια τα οποία δεν επισκέπτονται στο σχολείο τη σήμερα ημέρα. Αυτός δηλαδή ο πληθυσμός των 130 εκατομμυρίων είναι ο ίδιος ε, ο πληθυσμό με την δέκατη μεγαλύτερη ε, χώρα σε πληθυσμό στον κόσμο ή ανταποκρίνεται ε, στον πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Γαλλία μαζί. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει δηλαδή όλοι να συμβάλλουμε έτσι ώστε τα κορίτσια να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το δυναμικό του. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν δηλαδή του μηχανικού, του ιατρού και του ηγέτε του αύριο. Θα μπορούσαν να είναι εκείνε οι οποίε θα ε, ε, βρουν ε, θεραπείες για τις ασθένειές μας, να φέρουν μια επανάσταση στην τεχνολογία και να μας επιτρέψουν να διώσουμε πλήρως τη ζωή μας και εκείνες τις ζωές τους, όπως το κάνω εγώ, το κάνουμε εμείς και το, θα το κάνουν και οι κόρες σας. Θα πρέπει να προστατεύσουμε εκείνες τις, τις χώρε, στις φτωχότερες χώρες, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στην παιδεία για όλους. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα τολμηρό σχέδιο, αλλά χρειαζόμαστε και ευκολότερες πολιτικές, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την παιδεία για όλα ε, τα κορίτσια και προκειμένου να, ε, να υπάρχει ακριβώς η ε, οικονομική ανεξαρτησία για όλες τις γυναίκες, για όλα τα κορίτσια. Το 2015 οι ηγέτες του κόσμου είχαν αναλάβει από κοινού τη δέσμευση να τερματιστεί η Ένδια έως το 2030. Γνωρίζετε όλοι τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, ειδικότερα το στόχο υπαριθμών 4, που αναφέρει ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ε, την προσβάσιμη και ίση ε, εκπαίδευση και την παροχή ίσων ευκαιριών διαβίου για όλου. Εάν θέλουμε να επιτέχουμε αυτό το στόχο στο 2030, θα πρέπει να διπλασιάσουμε τι προσπάθειέ μα και τι επενδύσει μα αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε όλα τα κορίτσια έω το 2030 να επισκέπτονται το σχολείο. Ε, για να δώσουμε λοιπόν, να επιτύχουμε αυτήν την αυτεξουσιότητα για, τις, ε, για τα κόρτσα και τι γυναίκε ανά τον κόσμο, πρέπει να κάνουμε πολλά. Η παιδεία είναι το εφαλτήριο, αλλά θα πρέπει να κάνουμε και ε, παραπάνω πράγματα. Ειδικότερα αν θέλουμε να έχουν και περισσότερη οικονομική ε, Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως οι άντρες. Για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, δικαιώματα επί των γεών, ε, δυνατότητες απασχόλησης και πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας τις οποίες χρειάζονται. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ λίγο στον τομέα της υγείας ε, τα κορίτσια στις φτωχότερες χώρες έχουν πολύ υψηλότερο ε, κίνδυνο ασθενές και θανάτου κατά, την, κατά τον τοκετό. Η φίλη μου, για παράδειγμα, στο Καμερούν ε, ε, έχει πιθανότητα μία στις 180 να πεθάνει κατά το τοκετό, ενώ εγώ έχω μία πιθανότητα στις 4.900, δηλαδή 27 φορές ε, περισσότερο, περισσότερος κίνδυνος υπάρχει για τη φίλη μου στον Καμερούν. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε να μην υπάρχει τόσο μεγάλος κίνδυνος στο μέλλον. Και εγώ σε φοιτήτρια ιατρικής γνωρίζω ποιοι είναι οι κοινωνικοί παράγοντες, κοινωνικές ονιστώσεις που καθορίζουν την υγεία. Δηλαδή ένα κορίτσι το οποίο ε, ζει σε μια χώρα χωρίς υποστήριξη της οικογένειάς της θα έχει χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής και υψηλότερη πιθανότητα να πάσχει από σοβαρές ασθένειες ε, σε σύγκριση με ένα κορίτσι το οποίο ε, ζει σε μια ε, σε έναν ε, μεσαίου εισοδήματο ε, νοικοκυριό. Και βέβαια υπάρχει ε, και ε, ε, αυτό που λέμε ότι με βάση το ταχυδρομικό κώδικα μπορούμε να ξέρουμε το προσδόκιμο τη ζωή του καθενό. Και αυτό υπάρχει σε όλε τι χώρε. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε λοιπόν να χαθούν κι άλλε ζωέ κοριτσιών λόγω φτώχεια και λόγω ασθενειών ανά τον κόσμο. Εσεί λοιπόν ω Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο μπορείτε να μα βοηθήσετε προκειμένου να έχουμε αυξημένε επενδύσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα αυτά τα προγράμματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη 17,4 εκατομμυρίων επαγγελματιών υγείας ανά τον κόσμο. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει στο να κλείσει αυτό, να πληρωθεί αυτό το χάσμα και να βοηθήσει στο να έχουν όλα τα κορίτσια μια ε, πραγματικά μια ζωή στην οποία θα εκπληρώσουν τα όνειρά τους γιατί δεν ε, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ισότητα αν δεν είμαστε πραγματικά όλοι μας ίσοι. Σας ευχαριστώ. Ε, εμείς ευχαριστούμε λέει η Πρόεδρος. Τώρα, οι συνάδελφοι έχουν τον λόγο. Πρώτη, κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Thank you, Madam Chair. Uh, welcome. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ορίσατε. Και εκ μέρου ε, τη ομάδα δική συμφέροντα για τα δικαιώματα των κοριτσιών. Είμαι εντυπωσιασμένο από τα όσα μα είπατε και οι δυο σα. Έχουμε τώρα αυτή την εβδομάδα δράσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα κότσια. Θα μοιράσω τις συστάσεις σας τις οποίες μου δώσατε. Είναι πρακτικές, συγκεκριμένες. Μα είπατε για τις ε, τραγωδίες όσον αφορά του εξαναγκαστικούς γάμους, ε, τοκετούς, ε, ακροτηριασμούς. Να μην ξεχνούμε ότι πίσω από κάθε τέτοια περίπτωση υπάρχει μια τραγωδία, υπάρχει ο κίνδυνος ε, για το να καταστεί τραγωδία η ζωή μιας κοπέλας. Και είδαμε ότι υποστήριξη έχει αυτή η εβδομάδα μας ή έχουμε επίσης τις ε, συστάσεις προτεραιότητας που αντιστοιχούν ε, και στις δικές σας και οι δικές σας τις δικές μας. πολέμηση της βίας, πρόληψη της βίας, προστασία των θυμάτων της βίας, αύξηση συμμετοχής και ε, δεν θέλουμε να μιλάμε για σας, λέει το σύνθημα της εβδομάδας, θέλουμε ε, να μιλάμε με εσάς και με εσάς να συστάμε για σας. Χειραφέτης χρειάζεται, χειραφέτηση των ε, νέων γυναικών όσον αφορά την παιδεία και όσον αφορά την οικονομία. Όλα αυτά προσπαθούμε και είμαστε περήφανοι που είμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ο πιο μεγάλος δωρητής. η δράση πριν από έναν χρόνο. Τότε είχαμε τα μέτρα Τραμπ για τη, τη φήμωση και Έκοψε λοιπόν εκείνα τα κονδύλια. Εμείς προσπαθήσαμε να αντισταθμίζουμε αμέσως. Αναφέρατε την ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ήμουν σχετικά συνεισηγήτρια και με τους άλλους συναδέλφους προσπαθήσαμε να δούμε πώς θα αποσπάσουμε την υπογραφή των κρατών μελών για να προσχωρήσουν. Πάντως, Όπω είπατε, απομένουν πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Θα πρέπει να ενώσουμε τι δυνάμει μα, ώστε να ακυρωθεί και να εφαρμοστεί παντού αυτή η συμφωνία. Οπότε, η γάμη των ανηλίκων και όλοι, όλοι αυτοί οι εξαναγκασμοί θα πρέπει να ποινικοποιηθούν. Επίσης, πρόεδρε, ε, με αυτό το δίκτυο συνεργαζόμαστε στενά. Ναι. Και ήδη ξεκινήσαμε αυτή την εκστρατεία στις 6 Φεβρουαρίου. Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθούμε το θέμα να παραμείνει επί της τραπέζης. Πρέπει να προωθήσουμε τα ψηφίσματά μας. Ελπίζω θα τα λάβετε. Υπάρχει τόση πλειοψηφία εδώ για το έργο σας. για όλα αυτά τα προβλήματα, ε, τους πρόωρους γάμους, ε, ε, αναγκαστικές, αναγκαστικούς τοκετούς και νομίζω ότι όλοι οι προσβευτές αυτής της υπόθεσης όπως και εσείς κάνουν τρομερή δουλειά στη, στη βάση, στις κοινότητες, στη Πολύ πιο σημαντικό το τι κάνουμε εδώ. Οπότε είμαι και εγώ περήφανη που σε αυτή την εκστρατεία είμαι και εγώ πρέσβυρα και ασκώ αυτά, τα καθήκοντα ταπεινά. Σα ευχαριστούμε και πάλι. Εμεί ευχαριστούμε κύριε Κορατσαμπίλη, η πρόεδρο, κυρία Κοσλόφσκα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες Μισό λεπτό ρυθμίζουν ε, τα ακουστικά τους και την ε, κονσόλα της διερμηνίας οι δύο προσκεκλημένες. Τώρα με ακούτε, ακούτε τη μετάφραση. Λέει η κυρία Κοσλόσκα. Ε, Να τα powtórzę, Chciałabym się przyłączyć do e, słów pani poseł Anny Marii e, bildt. E, wszystkie komplementy, które płynęły w waszą stronę. κυρία να όλα αυτά τα συγχαρητήρια που είναι όλα δικαιολογημένα. Συμφωνώ σε όλα όσα είπε η κυρία Κορατσαμπίλη. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ, που καταβάλλατε την προσπάθεια να έρθετε στο Κοινοβούλιο και να μας πείτε, το, εσείς πώς βλέπετε αυτά τα θέματα, αυτά τα δικαιώματα των νέων γυναικών. Πώς βλέπετε εσείς τι θέματα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε αντιπροσωπείες από συναδελφού μας που πάνε στην Νέα τακτικά για αυτά τα θέματα. Πριν από δύο χρόνια πήγαμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα για τις ανήλικες γυναίκες. Είδαμε όμως ότι όσα και να συζητούμε, για τις γυναίκες που είναι το επίκεντρο της πολιτικής μας όσο και να συζητούμε θα πρέπει να ξεχνούμε λίγο ότι η ανισότητα αρχίζει πολύ νωρίς ξεκινά από την εφηβεία Άρα και εμεί θα πρέπει να λαμβάνουμε δράση για μια νωρίτερη φάση. Όχι όταν ενηλικιωθούν οι γυναίκες. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για τις ανήλικες γυναίκες, όχι μόνο τις ενήλικες. Άλλωστε, αν προστατεύσουμε τις ανήλικες γυναίκες, προστατεύουμε και τις μέλουσες ενήλικες. Βεβαίω έχουμε μια σειρά διαφορετικών προτεραιοτήτων ανάλογα με το που μένει κάθε νέα γυναίκα, Ευρώπη, Ασία ή αλλού. Βεβαίως είμαστε σε έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένο και ψηφιακό, η οποία μας αγγίζει όλους όπου και να ζούμε. Και αυτός ο ψηφιακός κόσμος μπορεί να αποτελέσει απειλή, μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικό αποκλεισμό. Από την άλλη όμως μεριά είναι και μια μεγάλη ευκαιρία γιατί χάρη στο ίντερνετ η απόσταση πια δεν έχει σημασία. Οπότε, ό,τι δεν ήταν στο παρελθόν δυνατό είναι τώρα. Οπότε μπορεί κανεί να κάνει μια σωροπρόντοτο στο Ιντερνετ η αποσταση πια δεν εχει σημασια οποτε οτι δεν ηταν στο παρελθον δυνατο ειναι τωρα οποτε μπορει κανει να κανει πια ενα στο ιντερνετ οπου και να βρίσκεται. Οπότε αυτό σα τονίζω το ότι αυτέ οι νέε τεχνολογίε, οι ψηφιακέ τεχνολογίε αποτελούν μια μεγάλη ευκαιρία ιδίω για τα κορίτσια, τις νέες γυναίκες που κατοικούν εκτός Ευρώπης αλλά και στην Ευρώπη. Και βεβαίως έχουμε διαφορές πολιτιστικές και κοινωνικές από χώρα σε χώρα. Πάντως εγώ σας ενθαρρύνω, σας προτρέπω, βοηθήστε μας να προωθήσουμε το θεματολογιό μας ούτως ώστε να καλύψει ο ψηφιακός κόσμος και τις νεαρές γυναίκες. Να μην υπάρχει χάσμα λόγω φίλου. Πολύ σημαντικές αυτές οι νέες τεχνολογίες. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να μπορούν όλες οι νέες γυναίκες να έχουν πρόσβαση. Χρειάζονται ανεξαρτησία και αυτονομία οι νέες γυναίκες πνευματικά με την παιδεία ε, οικονομικά με το να βρουν μια δουλειά για το Ιντερνετ βοηθάει σε αυτό. Και σας ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Κνιάσκα Κοσλόφσκα. Και τώρα θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να κάνετε τα καταληκτικά σας σχόλια, ενδεχομένως να έχετε και κάτι να προσθέσετε. Δεν ξέρω αν η φίλη μου από εδώ έχει κάτι να πει. Εγώ από πλευρά μου είμαι πολύ ευτυχής που μας υποδεχτήκατε εδώ σήμερα, που μας ακούσατε. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση για το έγγραφο το οποίο και υποβάλαμε, με χαρά θα τις απαντήσουμε είτε τώρα είτε και αργότερα. Και να μην ξεχνάτε ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί. Το κλειδί για να αποκτήσουν μεγαλύτερη ισχύ οι γυναίκες. Αυτά είχα να πω. Σύμφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το λόγο, που μας ακούσατε. Και φυσικά, αν έχετε ερωτήσεις και προς εμάς, ε, με χαρά θα τις απαντήσουμε. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα και που είσαστε τόσο νέες και τόσο δραστήριες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συστάσεις σας, γιατί εμείς οι πολιτικοί χρειαζόμαστε τις δικές σας συστάσεις και θα πρέπει να δράσουμε από κοινού. για να πετύχουμε αποτελέσματα αν θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σας ευχαριστώ και καλή μας τύχη. Runde. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διατάξη, το σημείο 11, η αποστολή στην Λιθουανία, στο EIGE. E. Αν δεν έχετε αντίρρηση, θεωρούμε ότι εγκρίνεται η έκθεση αυτή. Και περνάμε στο σημείο 11, αποστολή στην Εστονία. Δεν βλέπουμε να υπάρχουν ε, αντιρρήσεις. Εγκρίνεται λοιπόν και αυτή η έκθεση. Δεκατρία. Ε, σωματώσε τη διάσταση του φίλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, έχει ξεκινήσει, δεν έχει ακόμα καταφτάσει. Σε δύο-τρία λεπτά θα είναι εδώ. Να την περιμένουμε. Μέχρι να καταφτάσει η κυρία Μλίνλερ, Αγγέλικα Μλίνλερ.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 13 της ημερήσης διάταξης, ένταξη της διάταξης του φίλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η συγγήτρια είναι η κυρία Αγγέλικα Μλίναρ, εξέταση του σχεδίου έκθεσης. Να δώσω λοιπόν το λόγο στην συγγήτρια, την κυρία Μλίναρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρα, και θα ήθελα να διρετώ με μήπως χρειάζεται να περιμένουμε λίγο. Γιατί άλλο θα είναι μονόλογος η παρουσίαση αυτή. But you can you, I Ξεκινήστε. Ε, or maybe we can wait. Ξεκινήστε ή μήπως να χρειαστεί να περιμένουμε λίγο για την κυρία Αγνιέσκα Κοσλόφσκα που... Α, έφτασε και η Μαρία. Έφτασε η κυρία Νόχιλ. time we will wait a few minutes. Okay. Σα Thank you very much. Okay, dear colleagues. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συναδελφοί, αγαπητή Μαρία, αγαπητή Αγνιέσκα, να σας πω που βρισκόμαστε εν συντομία στο θέμα της ε, ενσωμάτωσης τη διάσταση του φίλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μόνιμη εισηγήτρια. Με χαρά θα σας παρουσιάσω το σχέδιο αυτή της διετούς ε, έκθεσης για το θέμα αυτό. Η τελευταία έκθεση, όπως ξέρετε, εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2016 και εξέτασα λοιπόν ποιες αλλαγές έχουν σημειωθεί έκτοτε. Καταρχάς όμως να σας δώσω μια επισκόπηση και μια παρουσίαση της γενικότερης αρχής τη έκθεση για την ενσωμάτωση τη διάσταση του φίλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπω ξέρετε, είναι ένα εργαλείο ευρέω αποδεκτό για να πετύχουμε καλύτερη ποιότητα, βάζοντα την διάσταση του φίλου στι προπαρασκευαστικέ δράσει, στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή και υλοποίηση των πολιτικών και των δαπανών και των σχετικών προγραμμάτων. Όλοι ξέρουμε ότι τελευταία αμφισβητείται ο όρος φίλο και άρα είναι ακόμα πιο σημαντικό από πολιτικής άποψη να καταλήξουμε σε σωστά αποτελέσματα. Είμαι πεπισμένη δε ότι το θέμα του φίλου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα της πολιτικής προκειμένου να προκύψει μια πολιτική συμπεριληπτική και σωστή ως προς το φύλλο. Εγώ λοιπόν ε, καλούμε να σας παρουσιάσω ποιες ήταν οι εξελίξεις και οι αλλαγές από τον Μάρτιο του 2016, 2,5 χρόνια, αλλά και οι πρακτικές ε, προτάσεις να κάνω για να βελτιωθεί περαιτέρω η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλλου. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω, φαντάζομαι, ότι ο πληθυσμός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντα αποτελείται και θα αποτελείται κατά το ίμιση από γυναίκε, αλλά δεν αποτυπώνεται αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη σύνθεση αυτού. 36,1% έχουμε ω ποσοστό ε, Ευρωπαίε ε, βουλευτές και αυτό συνεχίζει και στο Προεδρείο. 7 γυναίκε 13 άνδρες. Σε διοικητικό δε επίπεδο το ποσοστό των γυναικών σε ανώτατε θέσει είναι κάτω από 30% παρά το γεγονό ότι έχουμε πολύ πιο, υψη, πολύ πιο πολλές γυναίκες, αλλά όσο πιο, υψηλά, όσο πιο ψηλά κλιμάκια κινούμαστε, τόσο πιο πολλοί είναι άντρες. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί η δημοκρατική εκπροσώπηση των Ευρωπαίων πολιτών και ασφαλώς και η νομιμότητα των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή η πρεδική λοιπόν και επικριτική αξιολόγηση του που βρισκόμαστε είναι απαραίτητη και αυτό νομίζω ότι το πιστεύω όχι μόνο εγώ. Να ξεκινήσω με τα θετικά λοιπόν, γιατί καλωσορίζω ειλικρινά τη φιλόδοξη έκθεση του Δημήτρου Παπαδημούλη για την ε, ισότητα σε ό,τι αφορά τη διάσταση του φίλου στην ε, Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε ό,τι αφορά το 2016-2019 εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμένες περιορισμένα πρότυπα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ζητούν την ισότητα των φύλων και την ισότητα των ευκαιριών. Καλώ ορίζω και τι αναφερομένε κατευθυντήριε γραμμέ για τη χρήση ουδέτερη γλώσσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ω προ το φύλλο πάντα. Δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του τρέχοντο έτου. Και καλώ ορίζω το γεγονό ότι πιο πολλέ κοινοβουλευτικέ επιτροπέ έχουν εγκρίνει ένα σχέδιο δράση για την ένταξη τη διάσταση του φύλου. Το ακούσαμε και το πρωί. Πολλέ είναι οι προκλήσει που παραμένουν όμω, παρά το γεγονό ότι είμαστε 59% οι γυναίκε του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπροσωπούνται στα ανώτατα κλιμάκια, όπως σας είπα, του Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά τι προσλήψει. καλούμε λοιπόν τον Γενικό Γραμματέα και το Προέδριο να καταστήσουν υποχρεωτική τη συμπερίληψη των τριών άνω των αξιωματούχων με έναν εκπρόσωπο κάθε φύλου. Επίσης, επίσης θα πρέπει να προτιμάτε το υποεκπροσωπούμενο φύλο. Αυτό είναι ίσως σε πόθος, αλλά χωρίς να καταβάλουμε προσπάθεια δεν θα καταφέρουμε τίποτα ποτέ για να βελτιώσουμε την κατάσταση όσο έχει τώρα. Είναι επίση σημαντικό να συμπεριληφθεί και η κοινότητα ΛΟΑΔ στην έκθεση αυτή, γιατί η προβολή του προσωπικού ΛΟΑΔ είναι σχετικά χαμηλή. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προστατεύει τους εργαζομένους του από σεξουαλική παρενόχληση και βία. Καλό για πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Κοινοβουλίου στις 26 ε, Δεκάτου 2017 για την καταπολέμηση σεξουαλικής παρενόχλησης. Θέλουμε λοιπόν μεγαλύτερη ισότητα και στις πολιτικές ομάδες και στην γραμματεία του Κοινοβουλίου. Χρειάζεται λοιπόν μια αλλαγή νοτροπίας, μια αλλαγή στάσης, αν γίνει. Και τέλος, ε, θα υποβάλω τροπολογίες μεταξύ άλλων και για τα εξή θέματα. Να υπάρχει ειδική χρηματοδότηση για το φύλλο στον προπολογισμό, επίσης να υπάρχει σχετική εκπαίδευση των βουλευτών στην αρχή της θετίας τουλάχιστον, επαγγελματική εκπαίδευση για υποσυνείδητες πρακτικές παρενόχλησης και για να υπάρξει μια πιο καλή πρόθεση της έστασης του φίλου σε ό,τι αφορά τις προετοιμασίες ε, για τις επερχόμενες ευρωεκλογές ε, του χρόνου. Αυτά από πλευρά μου και να ακούσω με χαρά τα σχόλια των σκιεδών. Προσβλέπω και στις τροπολογίες σας και προσβλέπω άλλωστε και στην άριστη συνεργασία που χαρακτηρίζει την Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε την κυρία Αγγέλια, Αγγέλικα Μλίναρ. Να ακούσουμε τις σκιώδεις τώρα. Η Αγνιέσκα Κοσλόφσκα που εκπροσωπεί την κυρία Φάρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου του συναδέλφου, ο οποίο ε, χρειάστηκε να ε, παρευρεθεί στη συνεδρία τη άλλη επιτροπή αυτή τη στιγμή. Οπότε ε, μου άφησε ένα σημείωμα για να το διαβάσω. Και είναι το εξή. Αγγέλικα Μιλίνε, λοιπόν, απευθύνεται σε εσά. Θα ήθελα να σε συγχαρώ για μια ισορροπημένη ε, πρόταση σε ό,τι αφορά τη δουλειά που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι στιγμή σε ό,τι αφορά την ένταξη τη διάσταση του φύλου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει θετικά όλες τις το, προσπάθειες που έχουν γίνει και όπω αποτυπώνονται σε αυτή την έκθεση. Αυτό δηλαδή αποτελεί μια καλή αφετηρία για να συζητήσουμε τι πρωτοβουλίε, οι οποίε ε, τρέχουν αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο. Παρόλα αυτά, Παρ' όλα αυτά λοιπόν και κατά τη δική μου άποψη νομίζω πως θα πρέπει να λαφθούν υπόψη ε, ακόμα και κάποια ακόμα ζητήματα για παράδειγμα ως προς το πώς ε, η θα πρέπει να η έννοια του γάμου θα πρέπει να συσχετιστεί με αυτή την ένταξη τη διαστάση του φίλου. και ε, νομίζω πως κάποιες παράγραφοι επίσης θα πρέπει να διατυπωθούν με πιο σαφή τρόπο έτσι ώστε να μην υπάρξουν παρανοήσεις. Θα πρέπει να, είναι απόλυ... να είμαστε απόλυτα σαφείς ως προς το ποια είναι τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να υποστηρίξουμε την ένταξη τη διάσταση του φίλου στι ε, πολιτικέ. Ε, για παράδειγμα το roadmap, ο χάρτης πορεία δηλαδή για την αντιμετώπιση ε, της ε, πανενόχλησης σεξουαλικής ε, και άλλης, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευόμενους. Και επίσης θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε περαιτέρω τέτοια μέτρα. Επίσης θα πρέπει να εντοπίσουμε ακριβώς ε, ε, τις συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου θα πρέπει να παρέμβουμε και επίσης θα πρέπει να έχουμε ως στόχο πολύ συγκεκριμένα και πολύ απτά ε, αποτελέσματα. Για παράδειγμα, στην παράγραφο 12, εκεί όπου χαιρετίζουμε τα όσα έχουν γίνει σε επίπεδο αποφάσεων της, του, των Προέδρων, σε ό,τι αφορά δηλαδή την ενεργοποίηση τη Συμβουλευτική Επιτροπή, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των παραπούνων ε, για παρενόχληση, θα μπορούσε λοιπόν εδώ να γίνει μια προσθήκη η οποία θα προβλέπει μια σαφή εντολή απέναντι στην Επιτροπή. Επίση, ε, θα πρέπει να είμαστε σαφεί σε ό,τι αφορά τι επικείμενε ευρωεκλογέ. Ε, δηλαδή, στο πλαίσιο του αυτών των επικείμενων εκλογών μπορούμε να δημιουργήσουμε και έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε πιο Καλού ποιοτικά κανόνε για του ε, επόμενου οι οποίοι θα μας δεχθούν στο Κοινοβούλιο από το 2019 και μετά. Για να υπάρχει περισσότερη ισορροπία ανάμεσα στα δύο φύλλα. Ε, Καθώ είμαι και ο βασικό ε, συζητή σε ό,τι αφορά την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να αναφέρω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την ένταξη τη διάσταση του φύλου εδώ, στο δικό μα θεσμικό όργανο, στο Κοινοβούλιο. Εμεί θα πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα. Και θα κλείσω ε, συγχαίροντα για μία ακόμα φορά την συνάδελφο Αγγέλη Μινάρ και να πω ότι αναμένω με ενδιαφέρον τη στενή μα συνεργασία σε σχέση με αυτό το φάτελο προκειμένου να φτάσουμε σε, ένα, σε μια καλή έκθεση σε σχέση με αυτό το θέμα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο, ε, την κυρία Αγνέσκα Κοσλόφσκα και ευχαριστούμε και τον κύριο Φάρια, τον οποίο εκπροσωπήσατε. Δεν υπάρχουν άλλα μέλη που θέλουν να πάρουν το λόγο. Α, παρακαλώ. Ναι, να προσθέσω απλώς μια πρόταση ότι νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποτελέσουμε υπόδειγμα σε οτιδήποτε δηλαδή κάνουμε σε ό,τι αφορά τις συστάσεις ε, για την αλλαγή της νομοθεσίας απέναντι στους άλλους, απέναντι στα άλλα θεσμικά όργανα. Αν θέλουμε δηλαδή κάτι να αλλάξει, θα πρέπει εμείς να είμαστε υποδειγματικοί και τέλειοι σε ό,τι αφορά τη δική μας συμπεριφορά. Δεν, λοιπόν, ε, μπορεί να είναι ε, να, να κάνουμε δεκτό το γεγονό ότι υπάρχουν ακόμα διακρίσει ανάμεσα στα δύο φύλλα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξαλείψουμε αυτές τις διαφορές και να, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε να θεσπίσουμε ε, πιο αποτελεσματικούς κανόνες ε, στο μέλλον. Ευχαριστώ. Λέει Πρόεδρος, κυρία Φορέντζα, ως αστιός της ΕΓΚΟΕ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η εισηγήτρια ήμουν εγώ την τελευταία φορά και είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με την Αντζέλικα και με τι άλλε συναδέλφου και διαπιστώσαμε ότι είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. και μπορώ προσωπικά να σας πω ότι νομίζω πως ε, το έργο μας το ολοκληρώσαμε σε αυτή τη θητεία γιατί προσπαθήσαμε να αλλάξουμε την πολιτική του Κοινοβουλίου να υπάρχει ε, ακριβώς αυτή η συμπέριληψη τη διάσταση του φίλου στις πολιτικές του Κοινοβουλίου από το 2014 μέχρι τώρα και είπαμε τι γίνεται με αυτή την, την ουδετερότητα στις πολιτικές είπαμε να ε, μην εξετάζεται το φίλο σε, σε πολλές λειτουργίες τα κάναμε αυτά και σε σχέση με την Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορίου και έτσι όπως ξέρετε, προχωρήσαμε και σε μια έκθεση που είχε σημασία, που είχε σημαίνουν σχέση με τη διάσταση του φίλου στο διεθνές εμπόριο. Δικαιοσύνη για όλους θέλουμε. Δεν έχουν οικοδομήσει την ταυτότητά τους οι γυναίκες στο γυναικείο κίνημα επί τη βάση της χώρας προέλευσης, αλλά πρόκειται για αγώνες διεθνείς. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Και αυτό το mainstream και αυτή η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί δεν θέλουμε να περιστούμε μόνο στο θέμα το γυναικείο θέλουμε γενικότερα να επισημάνουμε τον κίνδυνο από τους νέους εθνικισμούς από ε, όλες αυτές τις ε, τάσεις που θα πρέπει κατηγορηματικά να καταγγείλουμε. Αυτό θα πρέπει να είναι η βάση, η αφετηρία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και έτσι θα αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που έχουν αναδυθεί. Θεωρώ ότι η εν λόγω έκθεση είναι πολύ σημαντική. Άλλο. Να αναγνωρίσουμε το πρώτο, το πόσο, πόσο σημαντικό είναι υπάρχουν οι χώροι, το περιθώριο για την ανέλυξη της γυναίκας. Να, πώς θα αποτελέσει κάτι το αποτελεσματικό, το mainstreaming. Στην Ιταλία υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχουν αυτοί οι χώροι, δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο. Δεν υπάρχουν αυτοί οι αναγνωρισμένοι, αυτά τα αναγνωρισμένα ε, μέρη. Και γι' αυτό και θα πρέπει να σταματήσει να υπάρχει σαν φρένο αυτός ο φόβος. Άρα σε αυτή την προοπτική της ισότητας των φύλων θα πρέπει να προχωρήσουμε και να βρίσκουμε τα μέσα για τις πολιτικές αυτές. Η δουλειά αυτή είναι πολύ σημαντική έτσι. Νομίζω ότι θα πιάσει τόπο η δουλειά όλων ημών όσο έγινε σε αυτή τη θητεία. Η ε, κυρία Νόχιλα Ευχαριστώ, Αγγέλικα. Θα ήθελα και εγώ να σε ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη πρότασή σου, που νομίζω πως θα οδηγήσει σε μια πολύ καλή έκθεση. Ε, ζητώ συγγνώμη που θα βάλω, έτσι θα χαλάσω λίγο όλα αυτά τα επενδυτικά σχόλια, αλλά εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι το θεσμικό όργανο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τις τοποθετήσεις της Επιτροπής ΦΑΜ. Δηλαδή είμαστε μια συμβουλευτική επιτροπή ουσιαστικά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ας μην έχουμε αυταπάτες και γιατί ε, συμβαίνει αυτό. Γιατί η πλειοψηφία δεν επιθυμεί ε, το να αναλάβουμε ένα πιο ε, θετικό ρόλο. Ε, δηλαδή όχι μόνο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά το σύνολο των πολιτών. Δηλαδή, εμεί μπορεί να λέμε ότι είναι πολύ σημαντικέ οι τοποθετήσει μα και θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη αλλά δεν συμφωνούν οι υπόλοιποι μαζί μας ε, και το βλέπουμε πώ ε, εκπροσωπείται έξωθεν ή από αλλού και οι διάφορε πολιτικέ ομάδε, εδώ. Δεν βλέπουμε δηλαδή του διάφορου ε, άντρε εδώ ψηλά αισθάμενου οι οποίοι συμμετέχουν στην Επιτροπή μα. Μόνο οι γυναίκε υπάρχουν εδώ. Άρα λοιπόν ουσιαστικά αυτό το κύρος, αυτό το ειδικό βάρος το οποίο θέλουμε να πείσουμε τον ένα στον άλλο μεταξύ μας ότι έχουμε δεν το έχουμε ως Επιτροπή. Και αν ε, δούμε αυτή η στρατηγική η οποία δεν μπόρεσε να περάσει για παράδειγμα κατά την έναρξη της βουλευτικής μας ε, θητείας ε, καταδεικνύουν το πού βρίσκονται τα πράγματα. Με μια τέτοια στρατηγική θα μπορούσαμε να είχαμε καταφέρει μια σειρά από τα πράγματα που αναφέρεις τώρα στην έκθεσή σου. Πολλά κράτη-μέλη ε, είχαν συμφωνήσει με, με αυτήν την ε, με αυτή τη στρατηγική 25 κράτη-μέλη από τα 28 κράτη-μέλη είχαν συμφωνήσει. Τα τρία ε, κράτη-μέλη έμειναν σε σιωπηρά. Ε, εκείνο λοιπόν η αντίρρηση ήρθε ουσιαστικά από πού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έδειξε ε, ιδιαίτερη. Ε, δεν, δεν στάθηκε στο πλευρό μας. και από την άλλη πλευρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκείνη ήταν που υπονόμευσε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή αποφάσισε να σιωπήσει και να μην προωθήσει μια στρατηγική. Άρα λοιπόν θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονό ότι η Αγγέλικα αναφέρει σε όλα αυτά τα σημεία και θα σε υποστηρίξω σε όλα τα σημεία που μπορώ, αλλά νομίζω πως η αλήθεια είναι ότι η πλειοψηφία ε, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σέβεται όσο θα έβρεπε τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτή είναι ε, αλήθεια και πραγματικά ε, έχω κουραστεί να, ε, να συζητώ ξανά και ξανά τα ίδια ζητήματα, να ε, συγχαίρουμε ε, τους εαυτούς μας για τις διάφορες λεπτομέρειες τις οποίες ε, διατυπώνουμε με διαφορετικό τρόπο, ενώ στην πραγματικότητα τα πράγματα παραμένουν όσο έχουν, δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα όσα λέμε και δυστυχώς τα πράγματα δεν βαίνουν καλώ λαμβάνοντας υπόψη και την άνοδο τη ακροδεξιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο στον Αγγέλη Καμλινάρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι που μου δώσατε την ε, δική σα άποψη και νομίζω ότι όλα όσα είπατε, όλοι σα είναι ακριβή και σωστά και αυτό που είπες Μαρία είναι κάτι το οποίο και εμένα με απασχολεί. Το λέω και ανοιχτά άλλωστε εκτός του Κοινοβουλίου ότι ουσιαστικά είμαστε μη νομοθετική επιτροπή και υπάρχει λόγο για αυτό. Αλλά να έχουμε υπόψη μα ότι ακόμα και όντας ε, μη νομοθετική επιτροπή, έχουμε έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Είναι πολύ μικρά τα βήματα της βελτίωσης, αλλά ουσιαστικά αγωνιζόμαστε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, για να μην ε, χειροτερεύσουν περαιτέρω τα πράγματα. Και αυτά που είπες Μαρία νομίζω ότι συνάδουν και με αυτά που είπε η Ελεονόρα πριν από λίγο. Χαίρομαι ιδιαίτερω. και για σένα Αγνιέσκα και τα σχόλιά σου γιατί δεν είναι καθόλου προφανή. <coughs> Χαίρομαι που είναι τόσο καλή η συνεργασία και νομίζω ότι θα πετύχουμε μια καλή έκθεση η οποία προφανώς δεν ταχθεί σε κάποιο πλαίσιο. Ιδάλλως ε, πολύ απλά θα την ε, κατέπνιγαν την έκτασή μας. Πολύ απλά θα πρέπει να εργαστούμε με τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και στο πολιτικό πλαίσιο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας στην παρούσα φάση. Συμφωνώ μαζί σου. Συνεργασία εθνικών δυνάμεων μαζί με πολύ συντηρητικές προσεγγίσεις διαφόρων εκκλησιών και φυσικά ένα από τους ε, Στόχου είναι η γυναίκα και το γυναικείο σώμα όλους ιδιαίτερο. Εν πάση περιπτώσει, προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σα και χαίρομαι ιδιαίτερω που σας έχω συναδέλφου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Αγγέλικα, λέει ο Πρόεδρος. Τροπολογίες. Μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Και τώρα να πάμε στο επόμενο ερώτημα. Στο επόμενο σημείο μάλλον. Μαρία Νόιτσελ. Point 14. Uh, Δημιουργία θέσπιση του προγράμματο, δικαιώματα και άξιε. Η κυρία Πιατικά είναι η συγκήτρια. Σχέδιο γνωμοδότηση, εξέταση αυτή. Η κυρία Κοσλόφσκα αντικαθιστά την κυρία Πιετικάινεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν μπορούσε να είναι εδώ η συνάδελφος. Βεβαίω ζητεί να την συγχωρήσουμε και μου άφησε κάποιες τι οποίε και θα σας διαβάσω. Αφορά αυτό το σχέδιο κανονισμού, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για αυτές τις αξίες. Το άρθρο 8 της Συνδίκης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θεωρεί ότι είναι στόχος της Ένωσης το να καθοριστούν αυτές οι αξίες που να πάσα δραστηριότητα. Η επίτευξη της ισότητας μεταξύ των φίλων είναι προς το συμφέρον μας και τέτοιες κοινωνίες θεωρούνται πιο δημοκρατικές και πιο σταθερές. Επίσης ε, η ισότητα οδηγεί και σε όφελος οικονομικό. Οπότε η συνολική πρόοδος από αυτού είναι πολύ αργή. Και έχουμε τους σχετικούς δείκτες του 2017 προς τούτο. Επίσης, έχουμε διάφορα επίπεδα δεσμένων διακρίσεων, έχουμε άνισες μεταχειρίσεις κατά των γυναικών και επίσης διάφορες μορφές βίας κατά των γυναικών. Αυτά όλα είναι κατά των βασικών δικαιωμάτων των γυναικών. Η, η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για, κατά της βίας αλλά και η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ακόμη δεν έχει κυρωθεί από όλα τα κρατημέλη. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να πετύχουμε την ισότητα των φύλων. Γι' αυτό το mainstreaming αυτή τη υπόθεση είναι πολύ σημαντικό. Άρα θα πρέπει να έχουμε κάποιους δείκτες, θα πρέπει να έχουμε κάποιον προπολογισμό, θα πρέπει να έχουμε το mainstreaming, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε ποιοτική λειτουργία των σχετικών προγραμμάτων. Πρέπει να καταπονομηθεί κάθε βία κατά γυναικών, ανηλίκων και ενηλίκων. Και θα πρέπει επομένως να προσέξουμε συγκεκριμένους τομείς με αυτό το πρόγραμμα για τις ε, αξίες. Και το Δάφνη επίσης. Οπότε η συμμετοχή των γυναικών θα πρέπει να εξασφαλίζεται στοχευμένα. Όποτε χρειάζεται. Μόνο με τέτοια προσπάθεια μπορούμε να πετύχουμε την ισότητα και τον τελικό στόχο. Το να μην υπάρχει αποκλεισμό, να μην υπάρχει βία και να υπάρχει ισότητα. Ευχαριστώ. Thank Εμείς ευχαριστούμε. Και τώρα, οι σκιώδες εισηγητές. Μαρία Νόιχελ, Σα Μαρία Ganz Σας ευχαριστώ και να διαβιβάσατε και στην εισηγήτρια και τους χειροτισμούς μου και τις ευχαριστίες μου. Είναι πολύ καλή η βάση και πιστεύω ότι πραγματικά όλα τα στοιχεία είναι εξαιρετικά. Να μην μας διχάζουν ως γυναίκες, σας παρακαλώ. Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι αναφέρεται και το θέμα των, θέμα των βιασμών των γυναίκων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το επίπεδο το οποίο αφορά όλες τις γυναίκες από όλες τις πολιτικές δυνάμεις το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να ζει χωρίς βία. Και γι' αυτό λοιπόν είναι αφεντικό. Το θα σας ανέφερε την αδελφό σας, θα καταθέσουμε τροπολογίες, αλλά επιτρέψτε μου να αναφέρω κάποια σημεία. Γενικά, καλωσορίζουμε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνεται στα δικαιώματα των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι θετικό ιδιαίτερα σε καιρούς όπου το θέμα των δικαιωμάτων ε, των γυναικών είναι πολύ επίκαιρο και πλήττονται τα δικαιώματα αυτά. Ιδιαίτερα λοιπόν τώρα είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει τις αρχές αυτές και τις αξίες αυτές, όχι μόνο με λόγια, με λόγια και πράξεις, όπως αναφέρεται και στη βίβλο Δεν φτάνει λοιπόν να τα γράφουμε όλα αυτά στο χαρτί. Είναι καλό λοιπόν το τι προωθούμε τις ιδέες αυτές. Τότε προκύπτουν συνέργειες. Πιστεύω ότι ως τώρα τα εφιστάμενα προγράμματα είναι καλά, αλλά όλα αυτά είναι θετικά μόνο εφόσον να εφροντίσουμε να μην υποτιμηθούν τα δικαιώματα των γυναικών. Τα προγράμματα λοιπόν να είναι πρακτικά, να έχουν καλές συνεργίες ως αποτέλεσμα, αλλά να μην ε, καταλήξουν να είναι όλα ίδια. Έχουμε λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή να επιστήσουμε στα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό θα πρέπει να μείνει στο επίκεντρο, να μην ε, καταλήξει να είναι δευτερεύουσα σημασία για τη χρηματοδότηση για τα επόμενα έξι χρόνια. Προφανώς η χρηματοδότηση είναι πιο χαμηλή από ότι σήμερα. Μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Brexit, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι α, πρόκειται για πάρα πολύ κακό σημάδι. Ένα κακό σημάδι γιατί εγώ έχω να σας πω όποτε μας χειροκροτούν αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν θέλουμε χειροκροτήματα, χρήματα θέλουμε, κονδύλια θέλουμε. Αφήστε τους επένους και τα χειροκροτήματα και άρα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε α, τα σωστά μέσα χρηματοδότησης και κυρίως ότι θα υπάρχει η μέγιστη αξιοποίηση των μέσων αυτών. Αυτό φυσικά δύσκολα ορίζεται. Να δούμε λοιπόν πού λαμβάνονται πολύ δύσκολες αποφάσεις από πλευράς των κρατών μελών, πού θα πρέπει να είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μέγιστη λοιπόν αξιοποίηση των κονδυλίων. Όσο πιο περιορισμένα είναι τα κονδύλια, τόσο πιο πολύ θα πρέπει να φροντίζουμε να υπάρχει καλή αξιοποίηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν την εισηγητρία που έβαλε μια καλή βάση και είμαστε όλε διατεθειμένε να συνεργαστούμε σωστά για να πετύχουμε το του δυνατό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Μαρία Λέι Πρόεδρο και τώρα από την Επιτροπή να ακούσουμε του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thanks uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια και τις ε, στιώδεις εισηγήτριες ε, για αυτήν την ε, γνωμοδότηση. Τη χαιρετίζουμε και τις προτάσεις που κάνετε σε αυτή και τις οποίες θεωρούμε σε έναν τρόπο να βελτιώσουμε το κείμενο. Νομίζω πως αντιλαμβανόμαστε εδώ ότι έχουμε κοινούς στόχους σε ό,τι αφορά ακριβώς ε, την σημασία και αυτού του προγράμματος και από ό,τι ε, διαπιστώνουμε υποστηρίζεται ε, τις προτάσεις που κάνουμε αλλά και τη δομή αυτής της έκθεσης. Για μας λοιπόν το λόγο πρόγραμμα είναι τα δικαιώματα δηλαδή και τι αξίε, πάρα πολύ σημαντικό και όπως ήδη αναφέρετε και εσείς θα θέλαμε ειδικότερα να δώσουμε έμφαση στο, στη διάσταση των αξιών. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε πολύ να ε, ε, να μην ε, μειώσουμε καθόλου την σημασία των σχετικών πεδίων πολιτικής τα οποία καλύπτουμε. Και γι' αυτό το λόγο η δομή που έχουμε επιλέξει δίνει ακριβώς την κατάλληλη έμφαση σε αυτούς τους τομείς και θίγει τα ζητήματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για αυτήν εδώ την Επιτροπή σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την ισότητα και την κατάβολαση των διακρίσεων, την ιδιότητα του πολίτη, το citizenship ε, και από εκεί και μετά αναμένουμε την ε, συνεργασία μαζί σας στις συνομιλίες και θεωρούμε ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε ένα πολύ ε, καλό και ισχυρό πρόγραμμα. Πρόεδρος, κυρία θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτές τις παρατηρήσεις και αυτές τις τοποθετήσεις. καθώς τα ακροδεξιά κόμματα ε, κερδίζουν όλο ένα και περισσότερο έδαφος, ε, είναι αναγκαίο να κάνουμε ένα διάλογο σε σχέση με τις αξίες. Ε, είναι δηλαδή ακόμα πιο σημαντικό να το κάνουμε τη σημερινή ημέρα. Πολύ συχνά, όταν συζητούμε τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακούγονται επιχειρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα χρήματα, δηλαδή με το ποια είναι τα χρήματα που λαμβάνουν ή δεν λαμβάνουν τα κράτη-μέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος της ε, και νομίζω πως ένα πρόγραμμα όπως αυτό το οποίο αναφέρεται στις αξίες ε, έχει νόημα. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 16 Οκτωβρίου. Περνάμε στο επόμενο σημείο τη σημερινή σα διάταξη, στο σημείο 15, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάση η συγγήτρια η κυρία Αγνέσκα Κοσλόφσκα. Εξέταση λοιπόν εδώ σχεδίου γνωμοδότηση. και δίνουμε λοιπόν το λόγο στην κυρία Κοσλόφσκα για να κάνει ω συγγήτρια την ε, παρουσίαση αυτής της, ε, του σχεδίου της νομοδότησης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus έχει πρικοδοτηθεί με περισσότερα ε, κονδύλια παρότι ε, το σύνολο εδώ του προϋπολογισμού σε ό,τι αφορά τα, την ε, πολιτική συνοχή έχει περικοπεί. Ο κύριος στόχος αυτού του ταμείου είναι οι άνθρωποι, η επένδυση στους ανθρώπους και κατά συνέπεια ο βασικός μου στόχος σε αυτή τη γνωμοδότηση ήταν να διασφαλίσω ότι αυτή η επένδυση στους ανθρώπους να γίνει λαμβάνοντας υπόψη και τη διάσταση του φύλου, ότι δηλαδή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ζητήματα της πρόβασης στην αγορά εργασία των γυναικών. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συνοδεύεται από την πρωτοβουλία για τους νέους, το πρόγραμμα για την υγεία και το ε, πρόγραμμα που καλύπτει ε, τον ε, ανάγκη συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων. Οπότε ο στόχος αυτού του προγράμματος και γενικότερα του κοινωνικού πυλώνα είναι να ε, ε, δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες και να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Νομίζω λοιπόν ε, και συμφωνούμε νομίζω όλοι σε αυτή την Επιτροπή ότι ο λόγος στόχος μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενίσχυση τη θέση των γενικών σε ό,τι αφορά τη μισθωτή εργασία και σε ό,τι αφορά την ισορροπία μεταξύ ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου τα όσα αναφέρθηκαν και στο σχετικό πακέτο για την ισορροπία μεταξύ ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου αναφέρουν ότι θα πρέπει ακριβώ να γίνουν περισσότερε επενδύσει σε, σε ό,τι αφορά τι σχετικέ υπηρεσίε που μπορούν να υποστηρίξουν τι γυναίκε. Άρα λοιπόν τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει να βοηθήσουν στην περισσότερη προσβασιμότητα των υφιστάμενων υπηρεσιών για τα εξαρτημέλη αυτά, ε, μέλη των οικογενειών των γυναικών, δηλαδή τέκνα και άλλου, έτσι ώστε να έχουν καλύτερη πρόσβαση οι γυναίκε στην αγορά εργασία. Ένα, μια ακόμα σημαντική διάσταση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού ε, Ταμείου σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης των γυναικών είναι η πρόσβαση σε ποιοτική και συμμετοχική ε, ε, παιδεία και συστήματα εκπαίδευση, ειδικότερα στον ε, ψηφιακό τομέα. Η μετάβαση δηλαδή στην ψηφιακή οικονομία και στη τεχνολογική αλλαγή μπορεί να λάβει χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο εάν γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επενδύσουμε εδώ περαιτέρω στι δεξιότητε των κοινοκών. Στο σχέδιο λοιπόν αυτό, καλό ε, για τη συμπερίληψη της διάστασης του φύλου ε, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ε, που αφορούν τις δεξιότητες στο πλαίσιο των χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Τέλος, η πρόταση για αυτό το ταμείο κάνει λόγο για υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων και μη άσκησης καμίας δραστηριότητα και επίσης αναφέρεται στην ανάγκη της βελτίωσης των επενδύσεων σε αυτό το τομέα. Υπάρχει μια μεγάλη διάσταση μεταξύ των δύο φύλων ε, σε ό,τι αφορά αυτούς τους νέους. Το 2017 για παράδειγμα το 21% των οικογενειακών από 22 έως 44 ε, ε, ήταν δηλαδή άτομα που ούτε εργάζονταν ούτε βρίσκονταν στην εκπαίδευση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών την ίδια περίοδο είναι το 13%. Οπότε θα ήθελα να καλέσω να ληφθεί υπόψη η διάσταση του φύλου κατά την, το σχεδιασμό του προγράμματο του Ταμείου δηλαδή, έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη και να εξασφαλιστεί ε, δραστηριότητα, δηλαδή είτε εκπαιδευτική είτε επαγγελματική, για αυτά τα άτομα τα οποία ακριβώ βρίσκονται εκτό εργασία και εκτό εκπαίδευση. Αναμένουμε ενδιαφέρον την συζήτηση που θα κάνουμε και τη συνεργασία με του στιώδει συζητητέ ε, σε σχέση με αυτήν την ε, σημαντική νομοθετική πρόταση. Σα ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Ανιέσκα. Και τώρα να δώσουμε το λόγο του σκιώδης εισηγητές. Εγώ είμαι μια σκιώδης ε, εισηγήτρια και θα πρέπει να σας πω τα εξή. πρωτα Πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω από καρδιά στην εισηγήτρια. Έχει επεξεργαστεί πάρα πολύ καλά αυτή την ε, τοποθέτηση. Βέβαια είναι η αρχική θέση που υπήρξε ε, και καλύπτει όμως ένα σωρό ζητήματα σχετικά με τις γυναίκες ίσως ε, σηκώνει κάποια βελτίωση το κείμενο και θεωρώ ότι η πρόταση της Αρμόδιας Επιτροπής θα πρέπει να κατατείνει στο να υπάρχει ένα ταμείο που να βοηθά τις γυναίκες που έχουν ανάγκη. Βλέπουμε ότι είναι στριμωγμένε οι γυναίκε, ιδίω οι πιο ηλικιωμένε, Άρα θα πρέπει να τονίσουμε ότι το εν λόγω ταμείο θα πρέπει να βοηθά περισσότερο τις ηλικιωμένε γυναίκες. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να επισημανθεί το εξής από το θέμα της παιδείας. Πρόκειται για την ισόβια εκπαίδευση, την ισόβια κατάρτιση. Μόνο έτσι θα αλλάξουν κάπως τα πράγματα. Εγώ είμαι πρόθυμη για συνεργασία και να επεξεργαστούμε κάποιες ε, τροπολογίες. Και έτσι το κείμενο γίνει ακόμα καλύτερο. Ευχαριστούμε και πάλι Ανίσκα. Mr. Pimenta is here and now I would like to give the floor. Ήρθε και ο κύριος Πιμέντα. Να ακούσουμε και την φωνή της Γκουέ από εσάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε μπόρεσα να ακούσω ένα τμήμα τη ε, παρέμβαση τη ε, εισηγήτρια σε σχέση λοιπόν με αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς, αλλά θεωρώ πως η συζήτηση σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες που μπορεί ε, να δώσει αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus σχετίζεται φυσικά και με τη ζήτηση που γίνεται σε ό,τι αφορά το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό ε, πλαίσιο. Γιατί ε, η σχετική πρόταση που έχει κάνει η Επιτροπή δείχνει να περιλαμβάνει σε ό,τι αφορά δηλαδή αυτό το πακέτο αν θέλετε των προτάσεων δείχνει λοιπόν να κινείται προς την κατεύθυνση της ε, περικοπής των κοντιλίων σε ό,τι αφορά και την πολιτική συνοχή αλλά και σε ό,τι αφορά τα ε, ταμεία τα οποία ε, προορίζονται για παρεμβάσεις κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα. Και αντιθέτως αυτή η δέσμη προτάσεων της Επιτροπής δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση άλλων, ε, ε, των, άλλων τομέων. Ε, δηλαδή ιδιαίτερη έμφαση σε ό,τι αφορά τον ε, στρατιωτικό και τον αμυντικό τομέα της Ευρώπης, για τον τομέα της ασφάλειας. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτών των ε, συζητήσεων, λοιπόν, εμείς δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ε, ξεχάσουμε, να παραγνωρίσουμε τη σημασία αυτών των ταμείων και, να συνεχίσουμε, και θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναφέρουμε τα δικά μας επιχειρήματα. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να συζητάμε τις δυνατότητες που μας παρέχουν αυτά τα είδη ταμείων συνοχής και ειδικότερα αυτό εδώ το ταμείο, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus και το πώς ακριβώς δηλαδή θα αξιοποιηθεί. Εμείς ε, έχουμε μια σειρά από τοποθετήσει ε, στι οποίε ήδη αναφέρεται η συγγήτρια και με τις οποίες δεν έχουμε κάποια διαφωνία, αλλά ε, υπάρχουν και μία σειρά από περαιτέρω ε, σημεία στα οποία θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή. Για παράδειγμα, στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν στις προτεραιότητες στο πλαίσιο δηλαδή των πολιτικών ανάπτυξή τους ε, ε, στα όσα προβλέπει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά του ζητήματα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια παρέκκληση από το γενικότερο όραμα, ε, το οποίο όπως σας είπα βέβαια ορίζεται και από το γενικότερο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και με βάση αυτό το νέο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο βλέπουμε ότι υπάρχουν περισσότερες αιρεσιμότητε πλέον, περισσότερε περισσότερες ε, προϋποθέσεις και βέβαια αυτό το ταμείο δεν θα αποτελέσει εξαίρεση ειδικότερα σε ό,τι αφορά δηλαδή στοιχεία μακροοικονομικής διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αλλά και άλλε αιρεσιμότητε. οι οποίες Ακριβώ είναι ε, και, και έχουν τελικά ως τελικό αποτέλεσμα την περικοπή των σχετικών κονδυλίων, ε, εν πάση περιπτώσει ε, επιτίθενται, περιορίζουν, περικόπτουν τα κοινωνικά δικαιώματα, οδηγώντα σε υποβάθμιση των δικαιωμάτων των γυναικών και οδηγώντα στην αύξηση της δυσμενούς διάκριση ει βάρος των γυναικών σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά του δικαιώματα. Ζητώ συγγνώμη για κινητό μου. Από την άλλη πλευρά, ο στόχος ε, του, αυτής της δέσμης προτάσεων είναι να δοθεί περισσότερη σημασία, περισσότερη εξουσία στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά την έγκριση αυτών των διαφορετικών ε, ταμείων. Ε, εμείς λοιπόν απορρίπτουμε αυτή τη νέα προσέγγιση, ε, δηλαδή των περισσότερων ρεσιμοτήτων αλλά και των περισσότερων εξουσιών σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και την έγκριση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί βέβαια όλα αυτά, αυτέ οι νέε προποθέσει, αυτή η νέα κατεύθυνση δεν θα διαφοροποιηθεί σε ό,τι αφορά αυτό εδώ το Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάσε. υπάρχει λοιπόν μια σειρά από πολιτικέ οι οποίε εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια ε, σε μια σειρά από κράτη-μέλη με βάση τις οποίες οι πολιτικές ε, ασκείται πραγματικά επίθεση απέναντι στα κοινωνικά δικαιώματα και φυσικά ε, στο πλαίσιο τη οποία τάση ε, ο αρνητικό αντίκτυπο είναι ακόμα μεγαλύτερο για τι γυναίκε. Άρα λοιπόν στο πλαίσιο και τη πολιτική ε, συνοχή, θα πρέπει να δούμε ποιε είναι ακριβώ αυτέ οι τάσει, ποιε είναι οι αιτίε για αυτέ τι τάσει και να ορίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει τα ίδια να ορίσουν ποιες είναι οι προτεραιότητες και οι ανάγκες τους σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική και από εκεί και μετά θα πρέπει να διασφαλιστεί ε, το πώς θα ορίζεται ο επιμερισμός των σχετικών ε, κονδυλίων ε, για αυτά τα κράτη-μέλη. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τεθούν στη δική μας έκθεση. Αλλά και όπως αναφέρθηκε και σε ένα σχέδιο γνωμοδότηση το οποίο θετήθηκε πριν από δύο-τρει εβδομάδε εδώ στην Επιτροπή μα. Ότι δηλαδή πέραν της, ε, ε άμεση, του άμεσου αντικτύπου σε ό,τι αφορά τη διάσταση του φύλου έχουμε και περαιτέρω δευτερεύουσες επιπτώσεις που και αυτές επηρεάζουν ε, την διάκριση ανάμεσα στα φύλλα. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι πολλές φορές η νομοθεσία η ευρωπαϊκή ε, δεν προβαίνει σε ε, διαφοροποίηση μεταξύ των δύο φύλων, αλλά τελικά η πρακτική εφαρμογή των λόγων νομικών πράξεων έχει διαφορετικό αντίκτυπο στα ε, διαφορετικά φύλλα. Και εδώ, σε ό,τι αφορά τι λόγω προτάσει, διαφορετικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τα δύο φύλλα σε σχέση με τα κοινωνικά του δικαιώματα. Εμείς λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε αυτή την πρόταση εδώ και αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία μόλις ε, έθιξα, τα οποία θεωρούμε πως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζωάπη Μέντα Λόπες, λέει πρόεδρος, και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Γιάνν Μπέγκρεν από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Yeah, thank you very... Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για τη δέσμευσή σας ό,τι αφορά την πρόταση αυτή για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Συν. Ενδεχομένω, από ό,τι κατάλαβα, να υπάρξουν περαιτέρω τροπολογίε. Είναι σημαντική η δουλειά αυτή για μα. Προσβλέπω και στη μελλοντική συνεργασία για το θέμα αυτό. Να πω δύο λόγια μόνο, επιτρέψτε μου, για αυτά που είπατε ως εισηγήτρης. Συμφωνούμε το ESF Plus, αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ, είναι μια φάση υποστήριξης ε, του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στο τμήμα επένδυσης σε ανθρώπους και όπως είπατε, βασική, βασικός στόχος είναι να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνέργειες για να σημειωθεί μεγαλύτερη επιτυχία από ότι με τα κεφάλαια. Είπατε ότι το ESF παρέχει βοήθεια στους πιο αδύναμους. Αναφέρθηκε και η πτυχή της ε, ένδυας. Έχουμε συμπεριλάβει το 25% κοινωνικής ε, συμπερίληψης και ένα ποσοστό για την στέρηση πρώτων υλών. Υπάρχουν λοιπόν ακόμα σε όλους τους τομείς ε, της ε, απασχόλησης κοινωνικής προστασίας και του καθεξής διαφορές ως προς τη διάσταση του φύλου. Αυτό το επισημάνατε εσείς. είχατε και το θέμα της συμφιλίωσης του οικογενειακού και του επαγγελματικού βίου. Όχι μόνο υπό νομοθετικούς όρους. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό και αυτό που είπατε για τους νέους. Παραμένει θέμα επικέντρωσης. Το ESF Plus παραμένει υπό κοινή διακυβέρνηση. Πολλά προγράμματα προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Εδώ λοιπόν επιστούμε προσοχή. Έχουν οριστεί τα επίπεδα. Αυτό που θέλετε να διευκρινίσετε δεν θεωρούμε ότι ήδη υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει με χαρά θα λάβουμε τις προτάσεις σας και σε ό,τι αφορά το παράρτημα των προτάσεων βλέπετε ότι έχουμε συλλογή δεδομένων φύλλο για όλους τους συμμετέχοντες προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει καλή παρακολούθηση της πρόοδου της διάστασης του φύλλου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Αγνιέσκα. Κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι της Επιτροπής, σας ευχαριστώ για όσα είπατε. Και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας πω ότι δεν συζητούμε γενικώ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτά απασχολούν την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Συζητούμε το κατά πώς θα πρέπει να αφιερώσει λιγότερους ή περισσότερους πόρους σε αυτή την υπόθεση η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς, ασχολούμαστε μόνο με το θέμα της όντας των δύο φύλων. Πάντως, είναι ξεκάθαρο ότι η ισότητα ανδρών γυναικών και γενικά ε, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα το πράγμα το πάνε καλύτερα είναι υπάρχει περισσότερος έλεγχος από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε ένα κύμα ευρωσκεπτικισμού που έχει φουσκώσει τώρα στην Ευρώπη. Σχετίζεται αυτό και με ε, κάτι, κάποια διστακτική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν θέλουμε δυνατή Ευρώπη, αν θέλουμε να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, αυτό θα δώσει περισσότερες πιθανότητες σε μια σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων για τα δικαιώματα των γυναικών. Χθες στην ε, Επιτροπή Προπολογισμών συζητήσαμε γενικώ για το μέλλον του προπολογισμού. Και είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο ταμείο για την θράξη της δημοκρατίας, ένα ταμείο να προστατεύει τα δικαιώματα των γυναικών και αυτό θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκού βεληνικούς. Μα έχουμε ε, για τις ε, επιμέρους χώρες κάποια ταμεία Ανατολή, Δύση, Νότο αλλά δεν υπάρχει τέτοιο ταμείο για γενικό χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κάτι που τώρα χρειάζεται, χρειάζεται πάρα πολύ. Μα, γι' αυτό σας λέω. Όσα λέμε, όσα προτείνουμε στην Επιτροπή των Προπολογισμών και οι τροπολογίες που έχουμε κατεβάσει θα πρέπει να υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επομένως να έχουμε κάποια ταμεία, κάποιους πόρους που να τους διαχειρίζεται ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι τα κράτη-μέλη. Έτσι θα έχουμε περισσότερη προστασία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών. tego funduszu. Tu chciałabym, żeby mnie przedstawiciel Komisji Europejskiej skorygował, ale... Τώρα, τι γίνεται από πλευρά ποσοτική. Α με γιορτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν κάνω λάθο. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια πρόταση περικοπή στον προπολογισμό να συρρυγνωθεί και το, το Ταμείο Συνοχή. Αλλά όμω το Γενικό Ταμείο πρόκειται να μεγαλώσει θα στο 27% του Ταμείου Συνοχής. Συμφωνώ με τα σχόλιά σας. Έχετε δίκιο. Η υπόθεση της φτώχειας των γυναικών είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να αναδειχθεί. Ιδίω για τις ηλικιωμένε γυναίκε είναι το θέμα σημαντικό. Γιατί έχουν μαζευτεί πολλέ ανισότητε σε όλη του τη ζωή. Και όλε αυτέ οι ανισότητε Επίσης ε, υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκε πληρώνονται λιγότερο. Κάνουν δουλειέ που πληρώνονται λιγότερο. Και εξελίσσονται στην ε, διαδρομή του πολύ λιγότερο από του άντρε. Έχουμε 40% κενό όσον αφορά τι συντάξει ανδρών γυναικών. Άρα, χρειάζεται πρόγραμμα ε, τέτοιο, σαν αυτό που συζητούμε τώρα, το ESF+. Plus. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί αυτή η παινία των ηλικιωμένων γυναικών. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί και ο κοινωνικό αποκλεισμό που είναι αποτέλεσμα αυτή τη φτώχεια. Επίση, Είπαμε να έχουμε περισσότερα προγράμματα για τι γυναίκε γιατί υποφέρουν περισσότερο οι γυναίκε από του άντρε από την ε, φτώχεια. Ε, άρα θα πρέπει να μπουν οι γυναίκε περισσότερο στου στόχου των προγραμμάτων. Ευχαριστούμε. 12 Οκτωβρίου έως τις 3 ε, ε, το μεσημέρι είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Περνάμε στο τελευταίο σημείο προσυζήτηση για σήμερα, 16 δηλαδή, πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικέ για την αντιμετώπιση των καρκίνων που προσβάλλουν τις γυναίκες και των σχετικών συνοσυρωτήτων. Η συγκήτρια είναι η κυρία Ντανιέλα Αγιούτου. Εξετάζουμε λοιπόν ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης αλλά και πρόταση ψηφίσματος. Ευχαριστούμε την Ντανιέλα που προσήλθε λίγο νωρίτερα εδώ στη συνεδρίασή μα και θα ήθελα να τη δώσω απευθεία το λόγο δεν συμμετέσχουν στην ε, συζήτηση προηγουμένως. Είμαι λίγο γρυπιασμένη σήμερα. Κοιτάξτε, όποιος έχει παρακολουθήσει τις εργασίες της Επιτροπής ξέρει πόσο με ενδιαφέρει το θέμα. Και είχαμε τελευταίους μήνες και κάποια ακρόαση. Σας λέω, είναι θέμα που με ενδιαφέρει, γιατί κατά τη γνώμη μου το θέμα δεν μας απασχολήσει αρκετά. Αυτές οι ιδιοτυπίες, τα χαρακτηριστικά αυτή τη ασθένεια, πόσο θίγουν τι γυναίκε. Τη natura psicologica, che non sempre vengono tenuti... Είναι και ψυχολογικέ οι πτυχέ του θέματος. Sì, è vero, bisogna considerare tutti i malati, però quando veniamo... Όλοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασθένειε, αλλά κυρίω οι γυναίκε. Και τελικά μπορούμε να τα καταφέρουμε να το ξεπεράσουμε και έχουμε τελικά και τις ε, πληγές, που δεν είναι πληγές της ε, εγχείρηση, αλλά είναι ψυχολογικές αυτές που χτυπάνε την ψυχή μας, την οντότητά μας ως γυναικών και χρειάζεται υποστήριξη ψυχολογική και κατά τη θεραπεία και κατόπιν όταν κανείς πρέπει να επιστρέψει ε, στη δουλειά, στην οικογένεια, στα παιδιά του. Δεν θα πρέπει να λείψει αυτή η υποστήριξη ψυχολογική. Επομένως, θα πρέπει είτε η Επίτροπη είτε το κράτος κάτι να κάνει. Να υπάρχει μια πολιτική, να υπάρχει μια πρικοδότηση και να υπάρχουν ε, εγγυήσεις πρώτα-πρώτα για πρόληψη, για παρακολούθηση, για πρόσβαση σε θεραπεία για όλες τις γυναίκες. Και αυτό να γίνεται σύντομα. Βέβαια, Έχουμε, έχουμε όλο ένα και περισσότερο υπηρεσίες ιατρικές που ασχολούνται με αυτά. Πάντως υπάρχει θέμα με την καθυστέρηση, με την αναμονή. Είναι υπερβολική. Και πολλές φορές το κόστος για κάποια γυναίκα της μεσαίας τάξης το κόστος είναι απαγορευτικό. Άρα είναι δύσκολο κανείς να έχει την σωστή διάγνωση. Να έχει τέλος τη διάγνωση που πρέπει. Τα έχει πει αυτά η Eurostat και επομένως αυτό είναι ένας φραγμός στο να καταφέρουμε να νικήσουμε το κακό. Να υπάρχει επομένως πρικοδότηση για αυτή την ψυχολογική υποστήριξη. να φροντίσουμε να πλαισοδούν οι γυναίκες από πλευράς αυτής της ε, ψυχολογικής υποστήριξης κατά την ασθένεια, όταν έχουμε την ιστερεκτομή, όλα αυτά είναι κροτηριασμό στην γυναίκα. Ε, άρα πρέπει να υπάρχει αυτή η υποστήριξη. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα πρέπει το κόστος να είναι κάτι που μπορούν να το φέρουν οι γυναίκες. Εδώ είναι θέμα κρατικής ενίσχυσης και βοήθειας. Έτσι διευκολύνονται τα πράγματα. Έτσι θα είμαστε περήφανοι για τη δουλειά μας, για το έργο μας. Και με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι θίγεται το ζήτημα. Και έλαμβανε υπόψη όλα όσα άκουσα από τους συναδέλφους για το κείμενο. Και περιμένω να ακούσω τις τυχόν παρατηρήσεις Ευχαριστούμε κυρία Ντανιέλα Αγιούτο και τώρα θα δώσω το λόγο στο σκύο Η κυρία Πετήρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγητρία για την εισαγωγή που έκανε και για την ε, μεγάλη της προσήλωση στο θέμα αυτό της καταπολέμησης του καρκίνου. Στο ΕΛΚ το θέμα αυτό είναι θέμα προτεραιότητας. Και γι' αυτό και υποβάλαμε προφορική ερώτηση και ψήφισμα. Πιστεύουμε ότι ο καρκίνος αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πρόβλημα που επηρεάζει όχι μόνο όσους πάσχουν, αποτελεί και κοινωνικό ζήτημα και οικογενειακό ζήτημα. Ξέρουμε ότι αυξάνεται δε ο αριθμός των ανθρώπων που πάσχουν από καρκίνο. Και τα κράτη-μέλη δεν μπορούν λοιπόν να το καταπολεμήσουν μόνο στο φαινόμενο. Θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να βελτιωθεί το κείμενο σε ό,τι αφορά το τμήμα που αναφέρεται στην έρευνα και στην έγκαιρη διάγνωση. Από εκεί ξεκινούν άλλωστε όλα. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ασθένειας και του ιδιωτικού βίου του κόσμου που πάσχει και των όσων ε, φροντίζουν τους ασθενείς. Να λάβουμε υπόψη τι γίνεται και με τις συνθήκες εργασίας. Να υπάρχει επίσης ε, ίδια προσέγγιση σε ό,τι αφορά τους ασθενείς άντρες ε, και τις ασθενείς γυναίκες, γιατί πρόκειται για την ίδια ασθένεια. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, στοιχεία για τη διάσταση του φίλου και επίσης να συμπεριλάβουμε και πιο σωστή άμα φροντίδα για τα άτομα τα οποία βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους. τις πρακτικές λοιπόν όσοι τις διαθέτουν. Ευχαριστώ σκιώδη σοσιαλιστών και δημοκρατών Σιλιάνα Μπορζάν αλλά μιας και δεν μπορεί να παραβρεθεί εδώ η κυρία Μπορζάν, να διαβάσω την παρέμβαση της κυρίας Μπορζάν για το ψήφισμα αυτό. Συμφωνεί η κυρία Μπορζάν με την εισηγήτρια στα βασικά θέματα του ψηφίσματος και της προφορικής ερώτησης. Θα ήθελε να υπογραμμίσει τη σημασία της πρόληψης και της έγκρισης διάγνωσης του καρκίνου. Θα ήθελε η Επιτροπή να λάβει δράση για να υποστηρίξει τις ε, ενέργειες της ΠΟΗ σε ό,τι αφορά τις πτυχές αυτές και να, ζητήσει, να ζητήσει μεγαλύτερη προσοχή για την έγκαιρη διάγνωση, ανείχνευση και τη βασική έγκαιρη διάγνωση του καρκινητών οθικών και του καρκίνου του τραχύλου. Τίφεται, λοιπόν και θέμα διαφορών σε ό,τι αφορά τη θνησιμότητα από τέτοιου καρκίνου στην Ανατολική και, Ευρωπαϊκή και Κεντρική Ευρώπη. Θέλει να καταπολεμηθούν οι διαφορέ μεταξύ των χωρών με σωστέ έγκαιρε και ευθυνέ διαδικασίες για την ανείχνευση του καρκίνου. Πιστεύει λοιπόν η κυρία Μπορσάν ότι θα πρέπει να υπάρξει μία σύνδεση με τα εθνικά και ευρωπαϊκά κέντρα για πιο σωστή υπαροχή πληροφόρησης μέσω σωστού ελέγχου και υπογραμμίζει ότι κάποια είδη καρκίνου σε κάποιες χώρες ε, δεν αναφέρονται στα σωστά ποσοστά γιατί είναι χαμηλότερο το επίπεδο της υγειονομικής περιθάλψης και πιστεύει η κυρία Πορζένα ότι στο θέμα αυτό θα πρέπει να μας επιτρέψει να βρούμε συμφωνίες. Θα πρέπει να δείξουμε έντονη αποφασιστικότητα για να βοηθήσουμε τις γυναίκες που πλήττονται από τον καρκίνο προκειμένου να ανακάμψουν. Και δεν βλέπω να ζητά κανεί άλλο το λόγο. Κύριε Ντανιέλη, έχετε κάτι να προσθέσετε. Όχι, όχι, όχι. Μόνο να ευχαριστήσω και την συνάδελφο και την ε, άλλη συνάδελφο που εκπροσωπεί την α, συνάδελφο που απουσιάζει. Πολύ πολύ χαίρομαι. Έτσι θα προχωρήσουμε το έγγραφο. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Πρόθεσμη για κατάθεση τροπολογιών είναι 15η Οκτωβρίου. Στα διάφορα. Τίποτα. Επόμενη συνεδρίαση τον Οκτώβριο στο Στρασβούργο στις 9. Στις Βρυξέλλες 8 Νοεμβρίου. 9 το Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις για την ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ και τη γραμματεία. Η Πρόεδρος ευγενικά ευχαριστεί και τους Δερμηνείς. Ευχαριστούμε όλους τους σύμβουλους. Καλό απόγευμα. Σας εύχομαι και καλή ξεκούραση.